από τους φιλελεύθερους και τις, από την Ενωμένη Αριστερά έχω αιτήματα για την ε, διορισμό στις ε, αντιπροσωπείες, στις αντιπροσωπείες. Αυτά ε, θα αναφέρουμε στα πρακτικά.